Επαναλαμβάνεται τώρα η συνεδρίαση του ε, Ολομέλειας ε, η οποία διακόπη στι 3 Μαου. Τα πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στην ε, Ολομέλεια τη 3η Μαου έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσει. Ωραία. Τα πρακτικά εγκρίνονται.